Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θέλετε να αρχίσουμε μήπως. Διότι είναι τρεις και τέταρτο Καθίστε λοιπόν στη θέση σας. Κυρία Κάσπαρη, κυρία Καζάκ. Thank Uh, το πρώτο μας θέμα, η έγκριση ημερήσιας διάταξης. Σχόλια, ερωτήσεις, ο κύριος Κάσπαρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από συνεννόηση με την γραμματεία της Επιτροπής, επιθυμώ να παρατηρήσω το εξής. Στην αυριανή ημερήσια διάταξη να συμπληρωθεί η Συμφωνία Συνεργασίας με τις χώρες ΙΖΑ. Έχει υποβληθεί το σχέδιο στο Κοινοβούλιο για σύμφωνη γνώμη και θα ήθελα αύριο να μπορέσει να γίνει μια συνομιλία με τους, τους πρεσβευτές των χωρών αυτών. Υπάρχει πρόταση, λοιπόν, έχουμε ένα συμπληρωματικό θέμα στη μερίσια διάταξη για την προσωρινή εταιρική σχέση με την Ανατολική Νοτιοφρική. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει έτσι. Πολύ καλά. Άρα με αυτή την αλλαγή, την προσθήκη μάλλον στη μερίσια διάταξη, μπορούμε να εγκρίνουμε τη μέση διατάξη. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο. Μας υπενθύμησε ο κύριος Κάσπερ ότι θα έχουμε έναν επιτετραμένο υπεύθυνο από τις χώρες αυτές για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Σημείο 2 της ημέρης της διάταξης. Έγκριση των πρακτικών. της συνεδρίασης της 3 η Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε ότι αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα έχουν εγκριθεί. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Όπως ξέρετε είμαστε συνδεδεμένοι ευθείας με το ίντερνετ. Εκτός από την συνεδρίαση που θα έχουμε και κλεισμένα των θυρών αργότερα, γιατί έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών, Προθεσμία καθάθεσης τροπολογιών για την ε, συμφωνία με την Κολομβία δεν μπορέσαμε για αυτό το φάκελο ε, των συνεντικών να καταθέσουμε, να ορίσουμε την ε, προθεσμία. Μαριδιδή, όπως ξέρετε, είναι εισηγήτη. Θα πρέπει τώρα να το καθορίσουμε διότι προβλέπεται η ψηφοφορία στις 6 Νοεμβρίου. Προτείνουμε λοιπόν προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ως τις 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Λίγη αυτή η προθεσμία, ελπίζω να το σημειώσατε. Εταιρική σχέση και συμφωνία με το Ιράκ. Ο Εμίλιο Μενέντες είναι εισηγητής για το θέμα αυτό και η Μαρία Βαβία απεφάσισε να παρουσιάσει το κείμενο Δεδομένου όμως ότι σταμάτησε κάποια στιγμή η διαδικασία, άλλαξαν τα μέλη της Επιτροπής η συγγήτρια ζητά μια νέα προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τις τροπολογι... Ε, προθεσμία τροπολογιών την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου το μεσημέρι και θα ψηφιστεί και πάλι η έκθεση αυτή της 6 Νοεμβρίου. Και τελικά, καλά νέα έχω να σας πω. Ίσχυση της γραμματείας μας, ο Πιεγό είναι ο νέος, νέο μέλος της ε, γραμματείας. Τον καλωσορίζουμε, δεδομένου ότι είμαστε μια πάρα πολύ φορτωμένη στη δουλειά επιτροπή. Καλωσορίσατε λοιπόν και καλή δουλειά. Σημείο 5. Α, όχι, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Σημείο 4. Η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. σε σχέση με την μικροοικονομική ε, βοήθεια έγινε η τρίτη τριμερής διαπραγμάτευση, η τρίτη τριμερής διαπραγμάτευση της 9 Σεπτεμβρίου, ο την Καζάκ θα μας παρουσιάσει συνοπτικά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, ήταν πάρα πολύ καρποφόρος η συνάντηση, διότι κατορθώσαμε να προοδεύσουμε σε πολλά θέματα, σε πολλά κείμενα που αφορούν το σχέδιο κανονισμού. Η Επιτροπή μας υποσχέθηκε να μας στείλει συμβιβαστικές προτάσεις για κάποια από τα σημαντικά θέματα που μας αφορούν, αλλά υπάρχουν ακόμη κύρια θέματα εκκρεμίως αναφορά τις ε, αποφάσεις που αφορούν τις κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις ή τις εφαρμοστικές πράξεις για το MFA. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη συνάντηση αυτή της τριμερούς ε, ε, ομάδας διαπραγμάτευσης θα ολοκληρώσουμε ε, τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να σας πω ότι όντως σημειώθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία συνάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Λοιπόν, για τους κανονισμούς που αφορούν ε, με τη Λατινική Αμερική και με την Κεντρική Αμερική τις ε, εμπορικές συμφωνίες υπήρχαν επίσης ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό ασφάλισης. Εγώ δεν μπόρεσα να προεδρεύσω. Θα ζητήσω από τους εισηγητές, τον Γιούργεν και τον Μπεντ Λάγκεν, να μας ενημερώσουν για τα αποτελέσματα. Προφανώς ελέγχθη ότι καταρχάς υπάρχει συμφωνία, αλλά μετά απέτυχαν τα πράγματα. Κύριε Λάγκε. Χθες συζητήσαμε, μάλλον ε, διεξήχθη ο τελικός τριμερής διάλογος ως αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου μπορέσαμε με κοινή προσπάθεια να, γίνουν, να επιτύχουμε να γίνουν δεκτές πολλές από τις τροπολογίες μας που είχαμε συζητήσει και μάλιστα πολύ περισσότερες από αυτές που αρχικά ήθελαν να δεχθούν ε, Συμβούλιο και Κομισιόν και ιδίω σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, προδιαγραφές, καθώς και την διαρκή παρακολούθηση της εξελίξεως των θεμάτων αυτών, καθώς επίσης και μια ρύθμιση του προβλήματος της μπανάνας, όπου επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα είναι διαφανής, η διαδικασία δηλαδή περιορισμού της διάθεσης στην αγορά, με την έννοια να προστατευτεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Συνολικά το αποτέλεσμα της προσπάθειας της ε, αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου είναι πολύ θετικό. Το μικρό πρόβλημα που μόλις ανέφερε ο Πρόεδρος είναι ότι διαπραγματευθήκαμε και συμφωνήσαμε και ότι το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεως καταγράφηκε από την Κομισιόν σε κείμενο. Τώρα υπάρχουν ορισμένα μικρά προβλήματα και δύο κάπως μεγαλύτερα, όπου η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου έχει απολύτω διαφορετική άποψη για το τι συμφωνήθηκε από αυτό που τελικώς περιλήφθη στο έγγραφο. Επομένως πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουμε ξανά σε διαπραγματεύσει με την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να είναι απόλυτα αξιόπιστα τα κείμενα σε ό,τι αφορά την απόδοση των όσων έχουμε ε, συμφωνήσει με τα δύο αυτά όργανα. Άλλα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο κ. Η κατάσταση των σχέσεων με την Κεντρική Αμερική είναι όλο και πιο δύσκολη και αποφασίσαμε εν τέλει αφού έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως με την Κολομβία και το Περού να βάλουμε ορισμένα πράγματα στο κείμενο και στο προήμιο αλλά και στο καθ' αυτό κείμενο κυρίως αυτό που έχει σχέση με το monitoring, τη διαρκή παρακολούθηση και επίσης την χρήση των ρητρών διαφύλαξης για την μπανάνα και ορισμένα άλλα προβλήματα που δεν θα τα αναφέρω τώρα. Αυτό που προτείνουμε εμείς να κάνουμε, άλλωστε ενημερώσαμε ήδη την Κομισιόν και το Συμβούλιο για το ποιο νομίζουμε εμείς ότι είναι το περιεχόμενο του συμβασμού, το κείμενό μας το έχουν ήδη, ξέρω ότι το ένα από τα δύο αυτά όργανα μας υποστηρίζει, το τι θα κάνει το άλλο δεν ξέρω. Υπάρχουν βέβαια κάποιες παρανοήσεις και για αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε αύριο τουλάχιστον ενδεικτικά επί του κειμένου μας που θεωρούμε εμείς ότι είναι το σωστό και θα ζητήσουμε τότε από τους εταίρους μας να δεχθούν και αυτοί τις διατυπώσεις μας. Σε ευχαριστώ. Σωστά αναφέρατε. Το θέμα της κεντρικής Αμερικής είναι ιδιάζων, διότι έχουμε πίεση από την Αφέτη ότι αποφάσισαν να μην αλλάξει το χρονοδιάγραμμά τους. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουμε εμείς να τηρήσουμε τους κανόνες μας και την αρχή μας, ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνενετική ψήφος, αν δεν υπάρχει για τον κανονισμό διαφύλαξη συμφωνία εκ των προτέρων, θα πρέπει να ψηφίσουν. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει θα είναι προσωρινή ψηφοφορία ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ώστε να ψηφίσει μετά από την δική μας ψηφοφορία για το κανονισμό διαφύλαξη ΑΦΕΤ. Ή λοιπόν θα ευρεθεί λύση σε αυτή την ε, ε, έλλειψη συμφωνίας μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει συμφωνηθεί, ή θα υπερψηφίσουμε αφήνοντας ε, τελικά την τελική απόφαση. Δεν ξέρω εάν κάποιος συμμερίζεται τη δική μου ερμηνεία ή θέλει να δώσει κάποια άλλη ερμηνεία. Όχι, βλέπω δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Νομίζω ότι είναι ο μόνος λογικός τρόπος να συνεχίσουμε. Well, The το καλύτερο θα ήταν να πείσουμε την Κομισιό να συμφωνήσει μαζί μας. ώστε να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Αλλά φαίνεται ότι είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να βρούμε μία εναλλακτική λύση και να ψηφίσουμε χωρίς να προδικάσουμε την τελική απόφαση που θα αφορά το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του ε, κανονισμού και η τελική ψηφοφορία θα λάβει χώρα βεβαίως τον Νοέμβριο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν συμφωνία... Έως αύριο θα ψηφίσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο που σας υποδεικνύω. Συμφωνία τα έχει καλώς. Πέντε. Δραστηριότητες της εποπτικής ομάδας. Αρχίζω με το Μερκοσούρ. Γιατί μου είπε ο κύριος Σούστα ότι πρέπει να φύγει, γιατί έχει άλλες δεσμεύσεις, κύριε Λούκα Σούστα. Πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ σύντομα να σας πω ότι το περιβάλλον των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ούτε αίσιο ούτε αισιόδοξο. Είχε ε, και λόγω των συμβάντων στην ε, Παραγουάη μετά από τη θεσμική κρίση που υπέστη η χώρα είχε αναβληθεί ο γύρος που προβλέπεται να οργανωθεί εκεί ε, βεβαίως ε, έγινε ε, ενεπλάκη πλήρως η Βενεζουέλα, αλλά έχουμε και εκεί είχαμε εκλογέ την προηγούμενη ε, εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά ε, χωρών ε, εισαγωγικών χωρών, χωρών που κάνουν εισαγωγέ. και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι και για μιλάμε για χώρες μεγάλες οι έχουν και σημαντικό ρόλο να παίξουν στην διεθνή ε, κατάσταση. Ε, απ' την άλλη πλευρά έχουμε μία στάση προστατευτική από πλευράς της Αργεντινής, όχι μόνο προς εμάς, αλλά προς όλες τις άλλες ε, χώρες. Βλέπουμε προστατευτικά μέτρα. Πρέπει να δούμε επίσης τι θα γίνει και η κατάσταση, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και με την Βραζιλία, που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για την Βραζιλία. 22 με 26 Οκτωβρίου θα λάβει χώρο ο επόμενος γύρος. Δεν θα είναι βέβαια γύρος ίσως με πολύ ε, πλήρη ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα έχει πιο πολύ πολιτική, πιο πολύ τεχνική ε, έτσι, υφή αλλά θα υπάρχουν ομάδες εργασίας όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά τα τελωνία, όσον αφορά τις τελωνιακές διευκολύνσεις προς το εμπόριο ε, και επίσης μια άλλη ομάδα εργασίας ε, για τις ε, επενδύσεις. Πάντως, πέρα από το ότι το περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, το γεγονός ότι θα υπάρξει νέος γύρος είναι οπωσδήποτε παρήγορο. Φυσικά θα πρέπει να καθοριστούν ε, περαιτέρω και κάποια πολιτικά ε, ζητήματα. Παραμένουν ανοιχτά κάποια θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία βεβαίως περιπλέκουν την κατάσταση. Όμως, τουλάχιστον είμαστε στην καλή θέση να πούμε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ε, και ε, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ο γύρος 22 ε, με 26 Οκτωβρίου, όταν θα έχουν αποσαφινιστεί κάποια σημεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την διαπραγμάτευση, ίσως θα μπορέσω και εγώ να είμαι πιο σαφής και να έχω λιγότερες επιφυλάξεις όσον αφορά την ίδια τη διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να προσθέσω κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε τον διαπραγματευτικό γύρο 22 26 Οκτωβρίου. Ε, Λούκα, έχει ε, λέει ο Πρόεδρο, ε, και μία συνάντηση με την Γενική Διεύθυνση Τρέβ. Τι έγινε εκεί? Ναι, ναι. Αυτές οι αξιολογήσεις που ανέφερα προκύπτουν και από τη χθεσινή συνάντηση για το ίδιο θέμα. Η άποψή τους είναι ότι κάποια από τα νομοθετικά ρυθμιστικά ζητήματα ε, έχουν συζητηθεί σε βάθος, έχει επέλθει συμφωνία ε, σε πολλά θέματα, υπάρχουν όμως ε, άλλα ζητήματα όπως ας πούμε οι εισαγωγές, οι δημόσιες προμήθειες κτλ. παραμένουν ακόμα ανοιχτέ. Κυρίως με την Αργεντινή υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα η Βραζιλία. Ίσως θα μπορούσε να συμφωνήσει να ξεκινήσει η διμερής ε, διαπραγματεύσεις ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα το κάνει γιατί οπωσδήποτε έτσι θα τεθεί ένα αμφιβόλο το σύνολο του διαπραγματευτικού πλαισίου με τις χώρες Μερκοσούρ. Επομένως, η οικία Γενική Διεύθυνση της, Γενική, της Κομισιόν είναι πάρα πολύ προσεκτική και εξαιρετικά επιφυλακτική όσον αφορά την πρόθεση και την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Πέραν αυτού βεβαίως, οπωσδήποτε θα συνεχίσουν ε, με κάθε τρόπο αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται, είτε πρόκειται για την πολιτική κατάσταση στην Παραγουάη, είτε πρόκειται για την ε, νέα είσοδο της Βενεζουέλας κτλ. δεν τους πτωούν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η εποπτική ομάδα, λέει ο πρόεδρος, είχε μια άλλη συνάντηση, μια τρίτη συνάντηση. Πίτερ, εσύ ήσουν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πω ότι σήμερα το πρωί έκανε σε ένα εξαιρετικό εργαστήριο πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, μήπως μπορείς να μας πεις δύο λόγια σχετικά με τις εντυπώσεις που αποκόμισε από αυτό το πρωινό Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφο μου δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τις διαπραγματεύσει ΣΥΤΑ. Η, τα καλά νέα, τα καλά νέα λέω, ότι η τελευταία εποπτική ομάδα για τον Καναδά συναντήθηκε Ε, και ο κύριος Πετρουτσιώνε, ο επικεφαλής ε, της διαπραγμάτευσης, είπε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και μάλλον θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία φέτος. Ε, επίσης ε, αναμένονται οι διαπραγματευτές τον Οκτώβρη και μην ξεχνούμε ότι εντωμεταξύ συνεχίζονται στις Βρυξέλλες οι εντατικές διαπραγματεύσεις έτσι ώστε ε, να υπάρξει η κατάλληλη συνεργασία και έτσι ώστε και ο Επίτροπος Δεγκούχτ να ε, αμβλύνει και τις τελευταίες δυσκολίες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ε, ζητήματα όπως ας πούμε ε, οι δημόσιες προμήθειες, διανοητική ιδιοκτησία, η ονομασία προέλευσης κτλ. είναι σημαντικά ζητήματα διαπραγμάτευσης. Να σας πω τώρα δύο λόγια σχετικά με ε, την συνάντηση που είχε ο κύριος Πετρουσιώνε, η τρίτη άτυπη στη σειρά που είχε με τους εκπροσώπους της ε, ομάδας μας, της, συγγνώμη, της Επιτροπής μας ε, σχετικά με το βόηο και το κρέας και το Χοιρινό ε, ε, υπήρξε συμφωνία. Παραμένουν τα πουλερικά και τα αυγά και κυρίως λόγω της καναδικής ε, πλευράς. Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ προσκολλημένος στα θέματα αυτά διότι πρόκειται για μια χώρα με ιδιαίτερα μεγάλες εξαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Όσον αφορά την ονομασία προέλευσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την κλωστοϊφαντουργία και όσον αφορά την αυτοκίνηση βιομηχανία, αλλά εκεί ο Καναδάς δείχνει να έχει μία πιο ε, άνετη κατά κάποιο τρόπο ε, στάση. Ε, αυτό που ε, με ενδιαφέρει είναι ε, να απαλληφθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα γεωργίας, γιατί μην ξεχνούμε ότι έρχονται και οι συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Όσον αφορά τώρα την, τις δημόσιες προμήθειες, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη ε, ε, πρόοδο, ε, γιατί οι συζητήσεις ξεπερνούν τις δεσμεύσεις του Καναδά στα πλαίσια της ΝΑΦΤΑ. Βεβαίω ε, σε περιπτώσει όπω είναι ας πούμε οι αστικέ συγκοινωνίε ε, ε, σε μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα εκεί υπάρχουν πολλές, πολλοί περιορισμοί. Από την άλλη πλευρά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία. Κυρίω όσον αφορά πατέντες, δηλαδή πρόβλημα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λόγω της ΑΚΤΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναθεωρήσει το κείμενό της, ε, κυρίως υπό το φως της ε, απόρριψης του κείμενου της ΑΚΤΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες ε, και τις ε, επενδύσεις και οι δύο πλευρές θέλουν να διασφαλιστεί ελεύθερη και ελεύθερη πρόσβαση καθώς επίσης και εισοδή και η αντιμετώπιση όλων των πλευρών. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υπάρχει ένας προστατευτισμός από πλευράς του Καναδά. Αλλά βεβαίως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν και θα καθοριστεί και το όριο ε, απελευθέρωσης. Ε, μην ξεχνούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, ε, αλλά συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Καναδάς απαιτεί οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν γίνουν σεβαστοί οι εργατικοί νόμοι. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή δεν μπορεί να ανοίξει ε, τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πριν από την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας λόγω των πολλών επικαλυπτωμένων θεμάτων. Ε, η, η έκβαση επομένως των συζητήσεων με τον Καναδά ε, έχουν επίπτωση και στις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς εξακολουθούμε να αξιολογούμε την κατάσταση αλλά βεβαίως όταν θα δούμε και τον πλήρη κατάλογο ε, των διαπραγματεύσεων τότε θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη άποψη. Πάντως ο κύριος Πετρουτσιώνε εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσει στο σύνολό τους είναι ε, ικανοποιητικέ και σιγά σιγά όλα τα κομμάτια μπαίνουν στην θέση τους. Ε, και ελπίζουμε ότι και πριν ε, και ότι γενικώ τα πράγματα θα πηγαίνουν αρκετά καλά η κυρία Σιλβάνα Κοχμαρή ε, συνεχίζει τις ε, προσπάθειές της και τις ε, διοργανώσεις που κάνει και αυτά και με την ευκαιρία να πω ότι η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ καλή. όλοι όσοι είναι σημαντικοί είχαν εκπροσώπους τους το Κοινοβούλιο, τη Κομισιόν, το Εμπόριο, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου και κάθε φορά που γίνεται συζήτηση κάτι καινούριο μαθαίνουμε, κάτι καινούριο ακούμε. Πάντως να πω ότι και η... να πω ότι γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν αισιόδοξο, γενικώ είμαστε... Είμαστε ευχαριστημένοι ε, από την κατάσταση και βλέπουμε ότι ε, ε, πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι καλά και ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και θα έχουν αίσιο τέλος. Πάντως αυτό είναι και το κλίμα του Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε και ενδεχομένως ε, θα καταλήξουμε κάπου σε κάποια συμφωνία η οποία κατά την άποψή μου θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και για τους δύο λαούς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολύ ε, θετικά αυτό που μας είπατε και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ε, καλό και θετικό για την ε, πολιτική μας νομιμότητα στα μάτια της Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά ε, σας επίσης το σημερινό εργαστήριο. Περνούμε στη Μόλδοβα τώρα. Η συντακτική συνεδρίαση έλαβε χώρα πρόσφατα. Κύριε Γιουνκλέρ, εσείς είστε ο εισηγητής, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως, την περασμένη εβδομάδα είχαμε την πρώτη συνεδρίαση της εποπτικής ομάδας για τις DCFTA για τις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μόλδοβας. Είχαμε μία λεπτομεριακή ε, ενημερωτική συνεδρίαση. Είχαμε τρεις τέτοιες συνεδριάσεις. Μας ενημέρωσε η Επιτροπή και μας ικανοποίησε ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στη Μολδαβία. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης η πρόσωπη της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να πω ότι ήδη μετά από τρεις γύρους διαπραγματεύσεων υπάρχουν πολλά κεφάλαια τα οποία έχουν προσωρινά κλείσει. Άρα έχουν συμφωνηθεί κάποια κείμενα προσωρινά. Βεβαίως έγινε και κλεισμένο το η συνεδρίαση. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν μόνο συναδέλφους αλλά μπορώ να σας δώσω περαιτέρω την εξή ενημέρωση. Στο δεύτερο μέρος συνεδρία ήταν και ο πρέσβης της Μολδαβίας, ο οποίος παρουσίασε τη θέση της κυβέρνησής του, της χώρας του, σε αυτή την συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και παρουσίασε και τις απόψεις των εταίρων μας εκ μέρους της Μολδαβίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ο τέταρτος γύρος συζητήσεων προβλέπεται στο τέλος Νοεμβρίου να λάβει η χώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Καλώς εχών των πραγμάτων λοιπόν και πάλι θα συναντηθούμε στην ομάδα εποπτείας ίσως γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, αν όχι του χρόνου στις αρχές της χρονιάς, τον Ιανουάριο και ζητήσαμε και από εκπροσώπους ε, των βιομηχανικών κύκλων να είναι παρόντες από τη Μολδαβία να έρθουν επίσης, ώστε να ακούσουμε όχι μόνο την άποψη των δημοκρατικών κύκλων αλλά και των επιχειρηματιών της χώρας αυτής. Μία τελευταία παρατήρηση δεν έχουν ορίσει σε αυτές τις ομάδες και όλες οι σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό ζητούμε όσοι δεν το έχουν κάνει να τους ορίσουν. για το θέμα αυτό. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με εσείς ότι οι πολιτικές ομάδες όντως πρέπει να ορίσουν και μέλη σε αυτή την εποπτική ομάδα από τη στιγμή που δημιουργείται κάθε εποπτική ομάδα στο να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τώρα, ο κύριος Ρόπισον για τη Ρωσία δεν είναι εδώ. Μπορώ να σας πω όμως, δεδομένου ότι τα έχω σημειώσει, ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αυτής της εποπτικής ομάδας και της Γενικής Διεύθυνσης Trade για να δούμε πώς προοδεύει το θέμα στο κεφάλαιο του εμπορίου. Και υποφελούμε τις ευκαιρίες για να σας πω ότι έμαθα ότι κάποιες συνεδριάσεις μονίμων εποπτικών ομάδων ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή ίσως. Δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα με κάποιες από τις δικές μας που συζητούμε σήμερα δηλαδή. Αυτό είναι λυπηρό πρέπει να πω. Πιστεύω ότι συγητές όλων αυτών των θεμάτων των υποπτικών ομάδων έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν χώρα και αυτές οι συνεδριάσεις. Και βεβαίως όταν οργανώνουν τις συνεδριάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είναι κάποιος αριθμός μελών παρόντα. Βεβαίως δεν μπορούν να παρίστανται παντού οι πάντες και πρέπει να συνεχίζουμε ακόμη γιατί να ξέρουμε ότι κάποια μέλη είναι απόντα. Και όταν έχουν συγκληθεί αυτές οι συνεδριάσεις, κατά την άποψή μου, πρέπει όντως να λαμβάνουν χώρα. Διότι δεν είναι αξιόπιστο εκ μέρους μας την τελευταία στιγμή να τις ε, ακυρώνουμε, διότι οι προσκεκλημένοι μας τι γνώμη θα συναντήσουν. Μου ελέγχθη ότι και 12 ώρες πριν ενημερώθηκαν οι εξωτερικοί επισκέπτες μας ότι ενώ είχαν ετοιμαστεί ακυρώνονται οι συνεδριάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσω σε όλους τους εισηγητές όλων αυτών των εποπτικών ομάδων τέτοιου είδους καταστάσεις να μην επαναλαμβάνονται. Να μην συμβαίνουν ούτως ή άλλως. 6. Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται σε εξαγωγές ξυλίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύκολος φάκελος από ό,τι γνωρίζω. Έχει σχέση με μία από τις διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΠΟΕ. Το Μάιο ήδη εμείς εδώ ψηφίσαμε και συστήσαμε στο Κοινοβούλιο να συνενέσει στην ε, ολοκλήρωση αυτής της συνωνίας. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν κατά κάποιο τρόπο είναι φαρμοστικός κανονισμός τεχνικής ε, φύσεως με στόχο να επιτρέψει στην Επιτροπή να μπορέσει με εκτελεστικές ε, ε, πράξεις να καθορίσει κάποιους δασμολογικούς συντελεστές. Η Προεδρία της Κύπρου με ενημέρωσε ότι ήδη έχουν εξετάσει την πρόταση αυτή και πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να καταθούν τροπολογίες. Πιστεύω λοιπόν με απλοποιημένη διαδικασία βάσει το άρθρο 46 ότι μπορούμε να εγκρίνουμε αυτό τον κανονισμό αλλά βεβαίως θέλω να ακούσω και την εισηγήτρια, την ε, Ινέζε Βάιντερε από το ΕΛΚ, στην οποία δίδω αμέσως το λόγο. Ε, thank you very much, ε, Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας υπενθυμίζω τα πιο σύντομα, τα πιο σημαντικά στοιχεία. Έχουμε πρώτα ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον για την προμήθεια ξυλίας από την Ευρώπη. Από την Ρωσία, συγγνώμη. Βεβαίως, για τις ποσοστώσεις που κατανέμονται στην Ευρώπη. Τρίτο, υπάρχει ένα πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες συμφωνίες μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας. Η διαδικασία για τις διαβουλέσεις και την επίλυση διαφορών προβλέπονται στη συμφωνία. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Όμως, στην έκθεση εφιστώ την προσοχή σας σε σημαντικά, σημαντικές ελλείψεις της απόφασης του Συμβουλίου, η οποία έχει περιλάβει διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει εφαρμοστικές πράξεις, ξεπερνώντας έτσι τα όρια του άρθρου 218 της συνθήκης της Λισαβόνας. Σημειώνω επίσης στην εκθεσή μου ότι εάν απόφαση του Συμβουλίου για Διεθνή Συμφωνία προβλέπει διατάξεις που κανονικά υπάγονται σε συναπόφαση, τότε αυτό σημαίνει ότι στερεί από το Κοινοβούλιο τις ε, αρμοδιότητες του περί συναπόφασης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να φροντίσει ώστε τέτοιε διατάξει να μην περιλαμβάνονται πλέον σε αποφάσει του Συμβουλίου για τέτοιου είδου συμφωνίε. Με ευχαρίστηση σας λέγω πάντως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθεια αυτή υπερίσχυσε, Συμβούλιο και Κομισιόν δέχτηκαν τα επιχειρήματά μας και θεωρούμε ότι η πρόταση κανονισμού υπό τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία μπορεί να προχωρήσει. Τώρα, όπως είπατε σωστά, η Επιτροπή έχει δώσει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή μας δηλαδή και γι' αυτό προτείνω να προχωρήσει με ταχύ ρυθμό και συμφωνώ μαζί σας ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε βάση απλουστευμένης διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Άρα σχόλια από άλλες πολιτικές ομάδες. Εσείς παρακαλώ. Κούτας. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Συμφωνώ με την εισηγήτρια σχετικά με την διαδικασία στο μέλλον και προσθέτω ότι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τέτοιες ποσοστώσεις άλλης χώρας και το υποστηρίζω και εγώ εν τέλει την απλουστευμένη διαδικασία. Συγγήτρια, και εγώ προσθέτω ότι αυτά που είπατε περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση. Ωραία, ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Ο κύριος Μικελάντζελο Μαργαρίτα. Δεν έχω και εγώ να προσθέσω τίποτα ιδιαίτερο στα όσα είπε η συγγήτρια και οι διάφοροι συναδελφοί σας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσει με ταχεία διαδικασία, διότι είναι κέριου ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία μας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις ποσοστώσεις ξυλίας το δυνατόν συντομότερο. Και αυτό προβλέπεται και με την προσωρινή ε, εκτελεστική πράξη. Όσο το, το συντομότερο, τόσο καλύτερα. Άλλο κανεί. Κύριε Σιγήτρια. Όχι. Όλα είναι ξεκάθαρα. Ωραία. Συμφωνήσαμε λοιπόν και με αυτό. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν απλουστευμένη διαδικασία. Τώρα. Θα μπορέσει να ψηφιστεί στην αυριανή μας συνεδρίαση. Στη δε ολομέρεια θα πάει σε ψηφοφορία τον Νοέμβρη. Και τώρα το υπαριθμό 7. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για θέματα τελωνιακής συνεργασίας που αναφέρονται στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι επιτροπή και η συγητής μας είναι ο κύριο Στάστινη, στον οποίο ξαναδίνω το λόγο. Είναι πολύ... Ε, είναι η ημέρα αυτή έχει πολλή δουλειά για μένα και για τα θέματα μου, δηλαδή ε, συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που μου δίνετε το λόγο για να μπορέσω να μιλήσω για την τελωνική συνεργασία, συμφωνία τελωνική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Στις 24 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής με τον Καναδά. Ε, για την ώρα αναμένουμε την υπογραφή. Εν τω μεταξύ έχουμε αναβάλει την προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών για τη συμφωνία αυτή μέχρι, αρχάς, μέχρι αρχών Νοεμβρίου. Μετά θα γίνει διαβίβαση στο Κοινοβούλιο και περί τις 26-27 Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην ε, δική μας Επιτροπή την συμφωνία αυτή. Η συμφωνία αυτή έχει τους εξής στόχους. Από το 1998 οι τελωνιακές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά βασίζονται σε συμφωνία τελωνιακής συνεργασίας και αμοιβαία αρρωγή σε τελωνιακά θέματα. Το 2005 ο Καναδάς επέδειξε ενδιαφέρον να συνεργαστεί στενότερα με την Ένωση για να εξασφαλιστεί ε, σε όλη την αλυσίδα ε, προμήθειας η ασφάλεια. Το σχέδιο συμφωνίας για την τελωνική συνεργασία ε, για θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Κομισιόν ήδη από τον Αύγουστο 2011. Στόχος της νέας συμφωνίας είναι η ενίσχυση θεμάτων τελωνιακής συνεργασίας για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού στο διεθνέ εμπόριο, στο διεθνές εμπόριο, και για παράδειγμα των εμπορευματοκιβατίων. Η συμφωνία αποτελεί τη νομική βάση για αυξημένη τελωνική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, για παράδειγμα για ελέγχους ασφάλειας, τεχνικές προδιαγραφές ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, στρατηγική συνεργασία σε θέματα επιθόρησης φορτηγών πλοίων, καθώς και συνεργασία σε διεθνή φόρουμ. Τα, επίσης ανοίγει το δρόμο η συμφωνία αυτή για, αμοιβαία, για συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώριση για την ασφάλεια της τελωνιακής συνεργασίας και μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου. Δηλαδή, οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αρχές του Καναδά συνεργάζονται. Από το 2008 υπάρχει πρόγραμμα το οποίο αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο της συνεργασίας αυτής και που επιτρέπει στα τελωνία να συγκεντρώνουν τις, τους ε, πόρους τους που βρίσκονται σε Σπάνιδα και έχουν πιστοποιηθεί 10.000 και πλέον ευρωπαϊκές εταιρείες ως αξιόπιστοι εμπορικοί εταίροι. Έχουν συμφωνήσει επίσης σε αμοιβή αναγνώριση με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία με τον Καναδά θα επιτρέψει να διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τέτοια συμφωνία και με τον Καναδά. Η, την συμφωνία θα διαχειρίζεται ένα κοινό όργανο, μια κοινή επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και θα μπορεί αυτή να λαμβάνει ε, εφαρμοστικές αποφάσεις και για την αμοιβαία αναγνώριση. Αυτή θα αποτελέσει την οροφή που θα καλύπτει όλη την τελωνιακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Η νέα συμφωνία θα βασιστεί επίσης στα βασικά στοιχεία του, συνόλου των προδιαγραφών της συμφωνίας WCO. Δεν έχει συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου απαιτείται για την ε, σύναψη της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Άλλες πολιτικές ομάδες? Όχι. Κομισιόν? ο κύριος Μιχαήλ Κασακράντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε σε αυτά που μόλις παρουσίασε ο εισηγητής. Βεβαίως είμαι θα ιδιαίτερως ευτυχής ε, για την θετική αξιολόγηση που έχει κάνει ο, ε, η, ο εισηγητής στην, στο προσχέδιο της εκθεσής του. Άλλωστε, όπως είπε και ο ίδιος ο εισηγητής, το Συμβούλιο την 24η Σεπτεμβρίου ενέκρινε ε, της, ε, την συμφωνία ή μάλλον ε, έδωσε άδεια έτσι ώστε να υπογραφεί η συμφωνία. Από μας πλευρά θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την έκθεσή του ε, και για το γεγονός ότι ε, έχει ενστερνιστεί τις προτάσεις μας. Ε, το σχέδιο σύστασης είναι στο, στα έγγραφά σας, λέει ο Πρόεδρος. Και ε, δίνει πράσινο φως λοιπόν ο εισηγητής στην σύσταση αυτή. told ε, λοιπόν, προσωρινό χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 8 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Ψήφος ε, στην Επιτροπή μας ε, το Νοέμβριο στη συνάντηση συνεδρία της Επιτροπής μας. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Είμαστε στο σημείο 8. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την ε, Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας βάσει της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι κάθε φορά που μπαίνει μια νέα χώρα στην Τελωνιακή ε, Ένωση πρέπει να ελεγχθούν ε, τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υπάρξει και μία αποζημίωση για τις τρίτες χώρες, ε, ε, προκειμένου ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και εδώ προέκυψε το, η τροποποίηση της συμφωνίας λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 24 Σεπτεμβρίου ε, έγινε η πρώτη συμφωνία. Όμως ακόμα δεν έχει σταλεί το κείμενο στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ε, αναβάλουμε το θέμα αυτό. Όμως, όμως, μπορώ να σας συστήσω την ε, έγκριση της συμφωνίας αυτής, ε, γιατί ε, υπάρχει ένα σχέδιο σύστασης στον φάκελό σας και επίσης προτείνομαι να γίνει να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και να υπάρξει και το σχετικό έγγραφο από το Συμβούλιο. Θέλει κανεί να πάρει το λόγο, αντιτίθεται κανεί σε οτιδήποτε. Όχι, φαίνεται ότι όλοι συμφωνείτε μαζί μου. Ο κύριος Κίνερα Κύριε Κριστόφ κύριε από την Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος ε, Κίνε δεν έφτασε ακόμα. Ε, θα είναι εδώ σε πέντε λεπτάκια. Πρόεδρος. Ναι, δεν μπορώ να σταματήσω όμως ε, την συνεδρίαση. Φαντάζομαι ότι και η Κομισιόν θα συμφωνήσει από τη στιγμή που αυτή διαπραγματεύτηκε την συμφωνία. μπορούμε να προχωρήσουμε εν ευθέτω χρόνο όταν θα έρθει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θα ακούσουμε την άποψή του και θα σας προτείνω και χρονοδιάγραμμα. Φτάνουμε στο σημείο 9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην γεωργία. πρόκειται για δεύτερη ανάγνωση για την οποία είμαι εισηγητής. Να σας υπενθυμίσω Να σας υπενθυμίσω πώς έχει η κατάσταση και ποιες ε, είναι οι διαφορές μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. σύμφωνα και με τις ε, αντίστοιχες ε, συμφωνίες με την Ουκρανία και την ε, Μολδαβία, προτείνουμε δύο ειδών τροπολογίες. Αυτές οι οποίες ήδη αναφέρονται στην πρώτη ανάγνωση, στη θέση δηλαδή βάση πρώτης ανάγνωσης στο, του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, αλλά και κάποιες άλλες κάποιες τροπολογίες, οι οποίες επανεισάγουμε στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, που δεν αλλάχτηκαν από το, από το Κοινοβούλιο, αλλά από το Συμβούλιο συμβουλευτικές λοιπόν διαδικασίες έτσι ώστε να υπογραφεί υπόμνημα ε, κατανόησης και ε, ε, στοιχεία τα οποία έχουν περιληφθεί στις προηγούμενες αντίστοιχες συμφωνίες τις οποίες ανέφερα και τις οποίες όμως ανέτεια το Συμβούλιο απέρριψε. τώρα υπάρχει αίτημα για ε, μονομερή ε, ε, αιτήματα όσον αφορά τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για την περίπτωση της γεωργίας. Εμείς προτιθέμεθα να συζητήσουμε με το Συμβούλιο έτσι ώστε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί η συνδρομή στην Γεωργία και το Κυργιζιστάν Ε, και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση των συναντήσεων που θα λάβει η χώρα την 16 Οκτωβρίου. Ε, όπως ε, ήθιστε έχουμε τέσσερις μήνες ε, για τη δεύτερη ανάγνωση, όμως το αργότερο στον, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα πρέπει να εγκρίνουμε το θέμα. Επομένως, 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Να σας πω επίσης ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σταθεροί πάνω στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να εγχειρηματοποιήσει τη διαδικασία επιτροπής έτσι ώστε να ελέγξει του, τις ε, εκτελεστικές εξουσίες ε, της ε, Κομισιόν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 strong on this. Και πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είναι δυνατόν να, να επιτρέψουμε στο Συμβούλιο να χρησιμοποιεί όπως θέλει την επιτροπολογία έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Η επιτροπολογία, η διαδικασία επιτροπής είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο και θέλει να δώσει στα κράτη-μέλη καθώς επίσης και στα εκτελεστικά όργανα της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης δυνατότητες να ε, ελέγξουν την, ε, τις εφαρμοστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί στην ουσία τα κράτη-μέλη δίνουν αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει εκ μέρους τους και επομένως πρέπει να ελέγχουν την ε, σωστή εκτέλεση των αποφάσεων. Ε, και επομένως η απόφαση για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κομισιόν υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου η διαδικασία εξέτασης ε, προϋποθέτει την δυνατότητα αρνησικηρίας από το Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο μπορεί να ελέγξει την ε, Επιτροπή και, εν βάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα ε, να, μόνο να ελέγξει και όχι να απαγορεύσει. Επομένως, είτε το Συμβούλιο θα πρέπει να δεχτεί αυτήν την ε, ε, ενδιάμεση λύση μέχρι ότου φτάσουμε σε συστημική, μάλλον διοργανική συμφωνία, βάσει και του κανονισμού πλαισίου που ε, συζητιέται και έχουμε εισηγητή για το θέμα αυτό τον κύριο Καζάκ, είτε θα πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι δεν θα υπάρξει καμία συμβολία. Επομένως, ξαναλέω, είμαστε πρόθυμοι, έτοιμοι να δεχτούμε κάποια διαδικασία επιτροπολογίας, ε, χωρίς όμως ε, την διαδικασία εξέτασης και ότι δεν θα αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές αντίστοιχες διαδικασίες. Έχω εξηγήσει ήδη στους ε, σκιώδες εισηγητές, μια και είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό, έχω εξηγήσει λέω τη θέση μου, η οποία είναι ότι θα και, και μάλλον το Κοινοβούλιο ε, έχει ενιαία θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, αλλά ήθελα να το πω και σε εσά στην ολομέλεια της Επιτροπής μας δηλαδή. Δεν θέλουμε ούτε να παγώσουμε το φάκελο αυτό, ούτε να τον σταματήσουμε, αντιθέτως μάλιστα. Θέλουμε να έχουμε ισορροπημένη θέση, μπορούμε να δεχτούμε την Επιτροπολογία υπό την προϋπόθεση ότι και το Συμβούλιο θα είναι αρκετά λογικό και δεν θα προσπαθήσει να μας επιβάλλει κάτι το οποίο εις το μέλλον δεν θα μπορούσαμε έτσι και να δεχτούμε. Παρατηρήσεις, Πολ Μέρφυ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το διαδικαστικό ζήτημα μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που λέτε, δηλαδή να επιμείνουμε στην ε, συμβουλευτική διαδικασία και όχι στην εξεταστική διαδικασία. Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή το Συμβούλιο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Αλλά φοβούμαι ότι ένα μνημόσυνο, μνημός, μνημόνιο συγγνώμη, ε, κατανόησης συνδεδεμένο και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βεβαίως είναι κάτι που μας προβληματίζει. Ναι, βεβαίω. Απλώ εμεί προσπαθούμε να βρούμε κάποια ενδιάμεση ε, λύση έτσι ώστε να χορηγηθεί η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία. Λοιπόν, ε, τώρα πρέπει να σας πω ότι είναι εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η κυρία Κιάρα Καπέλο είναι εδώ. Έρχεται η συνάδελφος, δεν έχει έρθει ακόμη. Έρχεται. I regret it. Κρίμα. Τέλος πάντων. Ξέχασα επίσης να σας πω ότι στο 8 ότι στην ε, συμφωνία είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, πίνακες Βουλγαρίας και Ρωμανίας προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 8 Νοεμβρίου του μεσημέρι. Τώρα, για το 9, για τη Γεωργία. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Okay. We have come to the end of first part of our meeting. Next. στο τέλος του πρώτου μέρους συνεδρίασής μας. Το επόμενο θέμα μας θα είναι οι συνεδρίες των συντονιστών. Διακόπτουμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Μπορούν να έρθουν στις 4,5 συντονιστές παρακαλώ. Παρακαλώ, είναι δυνατόν να είναι εδώ οι συντονιστές, να αρχίσουμε νωρίτερα. Πρέπει όλοι οι συντονιστές να συνενέσουν, έτσι, γιατί πρέπει όλοι να μπορέσουν να φτάσουν νωρίτερα. Αν είναι λοιπόν δυνατόν, Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν στις 4.30. Και όπως ξέρετε είναι και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση αυτή. Είναι παρόντες δηλαδή οι συντονιστές, η γραμματεία, η βοηθή του, η νομική υπηρεσία. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και κλεισμένο των θυρών. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρία.